Καλώς ορίσατε λοιπόν και πάλι αγαπητοί συνάδελφοι. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπα της εκπροσώπου εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εξ ονόματος της είπα της εκπροσώπου, ο Επίτροπος, ο κύριος Τηλιανίδης. Σας περιμένουμε, μην ανησυχείτε, είμαστε υπομονετικοί. Okay. On behalf representative... Εκ μέρους λοιπόν της υπάτης εκπροσώπου, ο Επίτροπος Χρήστος Ιλουρανίδης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε για να κάνω μια δήλωση εξ ονόματο της Αντιπροέδρου Φεντερίκα Μογκερίνη για την κατάσταση στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Μια κατάσταση η οποία είναι ρευστή. Θα γνωρίζετε όλοι τα τραγικά γεγονότα στο Κουμάνοβο, στα βόρεια της χώρας, κοντά στο Κωσυφοπέδιο και τη Σερβία εκφράσαμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες και τους φίλους των δολοφονηθέντων και των τραυματιών και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε τα γεγονότα αυτά ήταν πρωτίστως εγκληματική πράξη και δεν υπήρχε κάποια ο εθνοτικό κίνητρο. Γι' αυτό και ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει το γεγονός ότι όλα τα κόμματα ε, καταδίκασαν ε, ανεξάρτητα όλες αυτές τις δραστηριότητες. Ένα από τα κόμματα μάλιστα διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο για να βοηθήσει ε, τη διαπραγμάτευση μιας λύσης χωρίς ε, καμία καθυστέρηση. Θα ήθελα τώρα να περάσω στην πολιτική κρίση η οποία είναι μακρά και δεν θα πρέπει τα πρόσφατα γεγονότα να αποτρέψουν την προσοχή μας από το γεγονός αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένε εκκλήσεις για πολιτική λογοδοσία, για τα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτονται από τις υποκλοπές ε, των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων που δημοσιοποιεί ε, η αντιπολίτευση. Να επισημάνουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα παρετήθηκαν δύο υπουργοί και ο επικεφαλής της, ε, των μυστικών υπηρεσιών ανέκαθεν λέγαμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και συγκεκριμένο βήμα για πολιτική λογοδοσία και ότι ελπίζουμε ότι αυτές οι εξελίξεις θα συνεισφέρουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ε, στους ε, κρατικούς ε, θεσμούς. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθήσαμε και τις δύο διαδηλώσεις που έγιναν στα Σκόπια την Κυριακή και τη Δευτέρα είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ο λαός να εκφράσει ελεύθερα τις απόψεις του και στις δύο περιπτώσεις ε, υπήρχε ε, μια διαδήλωση η οποία έγινε ειρηνικά και υπήρχε κατάλληλος χειρισμός από όλες τις πλευρές, κάτι το οποίο θεωρείται πολύ σημαντικό. Ευθύ εξ αρχή, ε, όταν ξεκίνησε αυτή η πολιτική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε έκκληση για την αποκατάσταση του ομαλού πολιτικού διαλόγου μεταξύ ε, των βασικών κομμάτων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και καλωσορίζω το γεγονός ότι τρεις από τους συναδέλφους σας ε, ανταποκρίθηκαν ε, στο κάλεσμα του συναδέλφου μου του Γιωχάνες Χάν για να διευκολύνουμε το διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών και όπως θα γνωρίζετε είναι οι κύριοι Χάουιτ, Κούκαν και ε, Βάικελ μαζί με τον Επίτροπο Χάν. Ε, συναντήθηκαν εδώ στο Στρασβούργο εχθές και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα με τον Πρωθυπουργό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, τον κύριο Γκρουεύσκι και τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ε, τον κύριο Ζάεφ. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική συνάντηση είναι σαφές ότι και οι δύο πλευρές ε, λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους αυτή τη ε, διαδικασία διευκόλυνσης του διαλόγου. Έχουν γίνει βάθος συζητήσεις για τις ε, αποκλίνησες απόψεις και θα χρειαστεί φυσικά και περαιτέρω διάλογος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχαίρει τα κράτη για τη δέσμευσή τους για την ευρωπαϊκή διαδικασία και τις δημοκρατικές αρχές, καθώς επίσης και τη συμφωνία τους να βάλουν το συμφέρον της, χώρα ε, χώρας πρώτα απ' όλα. Προτρέπουμε λοιπόν όλε τι πλευρέ να συνεχίσουν τη δέσμευσή του υπό αυτό το πνεύμα και καλωσορίζουμε και την ε, διάθεσή του να συναντηθούν εκ νέου υπό την ε, σκέπη αυτής της διαδικασίας και καλωσορίζουμε επίσης και το γεγονός ότι τα τέσσερα ε, βασικά κόμματα είχαν ε, συνάντηση, συναντήθηκαν οι επικεφαλείς τους στις 14 και στις 18 Μαΐου και συμφώνησαν να ξανασυναντηθούν στις 26 Μαΐου σε μία απόπειρα να ε, εξεύρουν μία λύση. Διότι οι πολίτες της χώρας αυτής αξίζουν κάτι καλύτερο και όχι απλά μια πολιτική δήλωση και μια πολιτική σαστημότητα η οποία απλώς διαιωνίζεται και δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ε, του λαού. Γι' αυτό και ακριβώς καλούμε τους ηγέτες της χώρας ε, να αναλάβουν πολύ σοβαρά ε, υπόψη της ευθύνης τους και να βάλουν το συμφέρον τους κράτους πάνω από το συμφέρον των κομμάτων τους. Εκ παραλίλου η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει έκκληση προς τις ε, αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν όλους τους ισχυρισμούς ε, για πιθανές ε, παραβάσεις, ακόμα και τα όσα δημοσιεύτησαν για τις υποκλοπές, με ανεξάρτητο και διάφανο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει επίσης μία ομάδα νομικών εμπειρογνωμόνων για να εξετάσουν κάποια από τα συστημικά προβλήματα τα οποία είχε επισημάνει στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε εκφράσει την ανησυχία της, ε, ε, θέματα τα οποία προκύπτουν και από τις υποκλοπές. Αυτά τα συστήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου αυτή η υποψήφια χώρα να μπει και πάλι στο σωστό δρόμο όπως πρέπει. Ολοκληρώνοντας, η προσέγγιση μας συνολικά για αυτή την κρίση αποτελεί πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών, ε, χρησιμοποιώντας τα κοινά μας εργαλεία για να έχουμε ένα σαφές μήνυμα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν μέσω όλων αυτών συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά και με τους διεθνείς εταίρους μας επιτόπου προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Commissioner. Ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε του εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων από το ΕΛΚ. Ο Υπουργό Έντουαρτ Κούκαν. Δύο λεπτά. First Καταρχά, να συγχαρώ τον Επίτροπο <clears throat> γιατί ήταν πολύ καλή η ομιλία του, πολύ καλή η παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ, μας βοηθάει πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ελπίδα μου ότι η σημερινή, η τωρινή συζήτηση θα δείξει την υποστήριξη προς την Μακεδονία προς το λαό της και τις φιλοδοξίες του. Είναι σε καμπή η χώρα και αυτή η δύσκολη κατάσταση θα, έχει κρίσιμη σημασία και γι' αυτό πρέπει να εκφράσουμε την υποστήριξή μας. Ε, η Μακεδονία είναι αντιμέτωπη με μια σοβαρότατη πολιτική κρίση. Υπάρχουν σοβαρότερες προκλήσεις για την ασφάλεια και αυτό ε, θα ε, διατέρασε οποιοδήποτε πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη. Στο Κουμάνοβο με τα τελευταία περιστατικά βλέπουμε πόσο σοβαρή μπορεί να γίνει η κατάσταση. Η βαθύτατη πολιτική κρίση της χώρας είναι ε, ε, τέτοια που θα πρέπει να ε, δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή. Υπήρξε το σκάνδαλο για τις υποκλοπές που πρέπει να χειριστούν οι αρμόδιες αρχές. Ταυτόχρονα θα πρέπει οι πολιτικοί θύνοντες να ασχοληθούν με το θέμα της πολιτικής λογοδοσίας. Δεδομένης της κατάστασης ε, χρειάζεται διάλογος πολιτική ευθύνη και ε, πιο εντατικός πολιτικός ε, διάλογος. Αυτό το έτοιμο προέρχεται από όλες τις εθνοτικές ομάδες και από όλο το πολιτικό φάσμα. Είναι σοβαρότατες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα και θα πρέπει όλοι οι δημοκρατικοί μηχανισμοί να λειτουργήσουν αισίως. Μιλώ κυρίως για το Κοινοβούλιο που πρέπει να είναι η βασικότατη πλατφόρμα για δημοκρατικό ε, ε, διάλογο αλλά και έλεγχο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείξουν υπευθυνότητα και άνοιγμα όλοι οι πολιτικοί στη Μακεδονία αλλά και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ας μην ξεχνούμε παρακαλώ ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης είναι ένα από τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ε, υπερβούμε αυτήν την κρίση. Θα πρέπει να επανέλθει σε τροχιά η χώρα. Δέχεστε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Γλέζο. Κύριε Γλέζο, παρακαλώ. Θέλω να γνωρίσω τον συνάδελφο εάν γνωρίζει πότε ήρθαν οι σημερινοί κάτοικοι της ε, περιοχής αυτής την, στον τόπο αυτόν. Πότε ήρθαν ακριβώς τη χρονολογία. Ε, δεν ξέρω, εξηγήστε μου εσείς. Ο κύριος Χάουιτ από τις πλευράς των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Κύριε Πρόεδρε, ε, συναντηθήκαμε μια μέρα μετά τις ε, συζητήσεις διαμεσολάβησης. Τα αποτελέσματα είναι εμπιστευτικά, αλλά ξέρω ότι η συνάντηση αυτή κράτησε πολύ χθε το βράδυ, αντιμετώπισε δεπίμαχα θέματα και υπάρχει δέσμευση της χώρας ε, και όλων των πολιτικών δυνάμεων υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας. Ορισμένα σχόλια δεν αφορούν ε, μόνο τη συζήτηση αλλά τη χώρα. Πρώτα απ' όλα ε, δεν θα πρέπει να σταματήσει ε, η πολιτική απομόνωση αλλά πρέπει να προωθηθούν πρώτα απ' όλα δημοκρατικές διαπραγματεύσεις. Ποτέ δεν έχουμε υποστηρίξει εμείς ως ομάδα την, το μποϊκοτάρισμα το κοινοβουλευτικό θα πρέπει και ο κύριος Κούκαν να ε, μην ακολουθήσει την ε, ίδια γραμμή αυτών που θέλουν αυτό το μπλοκοτάρισμα. Κανείς δεν λέει ότι αυτές οι υποκλοπές είναι εντελώς κατασκευασμένες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια των πρέσβεων της Ένωσης για να υπάρξει λογοδοσία για όσα δεν έγιναν σωστά. Τέταρτον, πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις ε, στο δικαστικό σώμα, στην κοινωνία των πολιτών, στις εκλογικές διαδικασίες. Όλα αυτά είναι στο σχέδιο δράσης και στον υψηλού επίπεδου διάλογο. Οποιασδήποτε νέα δέσμευση ε, για προώθησή τους πρέπει να εξηγήσει γιατί είναι τώρα διαφορετική η κατάσταση. Κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο. Αλλά εφόσον ο επικεφαλής αντιπολίτευσης είναι στη φυλακή πρέπει αυτό να καταγγελθεί. Την προηγούμενη Κυριακή ήμουν στο Κουμάνοβο και είδα τα σπίτια τα οποία είχαν καεί και ήταν γεμάτα από τρύπε, από σφαίρες και στο εσωτερικό ε, δεν υπήρχε τίποτα. Ο, οι κάτοικοι τους έφυγαν τρέχοντας για να σώσουν τη ζωή τους και 18 την έχασαν. Ελπίζουμε αυτό να ήταν μεμονωμένο γεγονός και να μην υπάρξει επίδραση στις ε, διεθνωτικές σχέσεις. Αλλά πολλοί μου είπαν ότι θεωρούν ότι αυτό συνδέεται με την έλλειψη πολιτικής σταθερότητας. Η έλλειψη εμπιστοσύνη είναι από μόνη της επικίνδυνη. Έχω επανειλημμένα καταγγείλει ότι η έλλειψη συζητήσεων ε, ένταξης ε, μπορεί να επιφέρει επιστροφή των ε, συγκρούσεων. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε. Αυτό που συνέβη στο Κουμάνοβο και στη χώρα μπορεί να μην είναι άμεση ευθύνη της Ευρώπης, αλλά εάν εμείς θέλουμε τα πολιτικά κόμματα της χώρας να δράσουν υπεύθυνα όπως και εμείς, τότε μπορούν και εκείνοι να αναμένουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράει και εκείνη υπεύθυνα. Ευχαριστώ πολύ. Από πλευρά του ECR, ο Άγγελ Νταμπάσκι. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να επιμείνω στο εξής. Συμπάσχω με τις οικογένειες των θυμάτων. Θέλω επίσης να υποστηρίξω απόλυτα την ακαιρεότητα της φίλης αυτής χώρας. Είναι μια χώρα που βρίσκεται σε μία από τις χειρότερες πολιτικές κρίσεις. Πρέπει λοιπόν να δοθούν απαντήσεις στις κατηγορίες για διαφθορά. Να λοιπόν γιατί οι αρχές πρέπει να εξηγήσουν στην κοινή γνώμη τι ακριβώς έγινε. Επίσης Είμαι σαφώ υπέρ της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο εφόσον πάψει το μίσος και εφόσον τα θεμελιώδη δικαιώματα αναγνωρίζονται στη χώρα αυτή απέναντι στους Βουλγάρους στη Μακεδονία. Και να βασιζόμαστε στις σχέσεις καλής γετνίασης. Άκουσα πολύ προσεκτικά τα όσα είπατε κύριε Ζαμπάσκη. Δεν ξέρω αν πραγματικά πιστεύετε ότι η ΦΥΡΟΜ πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για σταθερότητα στα Βαλκάνια, ότι πρέπει να μπει στον ΝΑΤΟ, μπορεί να είναι καλό για σας, για τη χώρα σας, για τις γείτονες χώρες, ίσως και για την Ελλάδα, να βοηθήσουμε την Μακεδονία στον ε, δρόμο που παίρνει ως φίλη της. Και ξέρετε εγώ μιλάω για δημοκρατία της Μακεδονίας και όχι για τέος δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. Ε, Αν ε, κατάλαβα καλά την ερώτηση, θέλω να σας πω ότι όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κριτήρια ε, τον σεβασμό τους, νομίζω ότι αυτό αυτό είναι η μόνη δυνατότητα για αυτό το κράτος για να διατηρήσει την εδαφική του καιρότητα, βεβαίως τηρώντας τα ευρωπαϊκά κριτήρια και επιπλέον ε, τηρώντας ε, τις ρήτρε της ε, Σύμβασης Καλής Γειτονίας. Εκ μέρους των ο κύριος Βάγγελ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Θέλω κι εγώ να σας ευχαριστήσω για τα ξέρετε λόγια σας και για την τόσο σαφή εισαγωγή που κάνατε στη συζήτηση αυτή. Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε τη Μακεδονία με μεγάλη πλειοψηφία ως χώρα που θέλουμε να δούμε μεταξύ μας την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζοντας βέβαια ότι η χώρα αυτή πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την ένταξή της. Αν δεν είμαστε εκεί ακόμα, αυτό οφείλεται στη σύγκρουση αυτή την ανόητη για το όνομα αυτής της χώρας. Η σημερινή συζήτηση δυστυχώς δεν έχει να κάνει μόνο με την ανανέωση της θετικής άποψης που έχουμε για την πρόοδο της Μακεδονίας ως υποψήφια χώρα, αλλά η πολιτική κρίση και τα τραγικά γεγονότα του Κομάνοβο αποτελούν μια προειδοποίηση για τα εθνικά και εσωτερικά προβλήματα στη χώρα αυτή της Νότιας Ευρώπης. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις απειλές του Ισλαμικού εθνικισμού και την στάση της Ρωσίας. Η κατάσταση στη Μακεδονία απαιτεί περισσότερη κατανόηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει επίση να βρούμε κάποιο συμβασμό για την ονομασία αυτή τη χώρα και να ανοίξουν τελικά οι διαπραγματεύσει με την Μακεδονία. Λέω Πρέπει να στηρίξουμε τη Μακεδονία στον δρόμο που έχει επιλάξει για να ενταχθεί και στο ΝΑΤΟ. Όσον αφορά τώρα τις σχέσεις της με την Ελλάδα, την γείτονα χώρα της, η χώρα αυτή που έχει όλη μας την υποστήριξη πρέπει να ξεχάσει πολύ στενά συμφέροντα για την ονομασία της γειτονάς χώρας. Επιπλέον, ο Αλβανός Πρωθυπουργό απείλησε ότι θα μπλοκάρει τις προσπάθειες της Μακεδονίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι η πολιτική της Μακεδονίας που είναι υπεύθυνη για την πολιτική αυτή εσωτερική κρίση πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για το μέλλον το ευρωατλαντικό αυτής της χώρας. Με τον Επίτροπο για τη Διεύρυνση, τον κύριο Χάν, έχουμε ήδη δεχτεί πολλά. From, uh, Mr. Υπάρχει μπλε κάρτα από τον κύριο Πετίδιο. Ναι, βεβαίως τη δέχομαι. Ευχαρίστω. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Πετίδιο. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, άκουσα με πολύ προσοχή την τοποθέτησή σας και διαπίστωσα ότι μόλις τώρα διαπράξατε μια απρέπεια. Χαρακτηρίσατε ως ανόητη τη διαμάχη της Ελλάδος με τα Σκόπια για το θέμα του ονόματος. Και ρωτώ, εάν αυτό συνέβαινε στη δική σας χώρα, εάν τα Σκόπια είχαν εκφράσει επεκτατικές βλέψεις για τη δική σας χώρα, εάν καθιονδήποτε τρόπο έφυγαν τη δική σας χώρα. Θα, είσατε, θα είσαστε τόσο άνετος για να πείτε αυτά τα οποία είπατε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Θέλω να σας πω ότι στην εποχή μας όταν είχαμε πολύ πιο σημαντικά θέματα Νομίζω ότι το πρόβλημα αυτό μοιάζει με τεχνητό, μια τεχνητή σύγκρουση και θα πρέπει να σταματήσει. Δεν έχει νόημα πραγματικά. Ευχαριστώ. GUE Group, uh, Deputy Sofia Sakorafa, one minute. Η κυρία Σακοράφα, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, μόλις πριν από δύο μήνες στη συζήτηση της ετήσιας έκθεσης πρόοδου για τη ΦΥΡΟΜ είχα τονίσει ότι η πολιτική της επιβράβευσης όλων αυτών των αρνητικών που συνθέτουν τη σημερινή κατάσταση της χώρας μόνο ανασταλτικά θα μπορούσε να λειτουργήσει για την πρόοδό της. Δυστυχώς τα γεγονότα στο Κουμάνοβο με επιβεβαίωσαν με τον τραγικότερο τρόπο. Στη γειτονική μας χώρα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία κράτους δικαίου, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την εφαρμογή της Διεθνωτικής συμφωνίας της αχρίδας τον σεβασμό της αρχής της καλής γειτονίας και το έλλειμμα της δημοκρατίας στη χώρα. σε αυτά ακριβώς οφείλουμε σαν ευρωπαϊκή ένωση να εστιάσουμε την προσοχή μας όλες οι άλλες αιτιάσεις περί εξωτερικών ευθυνών δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να εξοραίζουν την πραγματικότητα να διαιωνίζουν αυτή την τραγική κατάσταση και να βαθαίνουν φυσικά την κρίση. η συνέχιση αυτής της τακτικής και της πολιτικής κύριοι συνάδελφοι πέρα από όλα τα άλλα συνιστά ευθεία υπονόμευση των αρχών της ευρωπαϊκής ένωσης ας μην το ξεχνάμε αυτό και αποτρέπει οποιαδήποτε δυνατότητα προόδου και εξέλιξη της χώρας που λέγεται fyrom. Ευχαριστώ. Ο... Deputy Tamas Εκ μέρους των Πρασίνων ο κ. Μάζεριτς. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι Πράσινοι συμφωνούμε πλήρως με τους υπόλοιπους συναδέλφους που λένε ότι η κατάσταση στην Μακεδονία είναι ε, σοβαρή και εγκυμώνει περαιτέρω κινδύνους. Η κρίση τις ρίζες της ε, είναι περιφερειακή και, και βέβαια πολύ εσωτερική. Όμως δεν μας εκπλήσει, δεδομένου ότι η χώρα περιμένει 10 χρόνια για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μας εκπλήσει ότι χάνει την πολιτική της ισορροπία. Η Μακεδόνια, η Μακεδονία έγινε ο πρίγκιπας της ο, ο σε ό,τι αφορά την ένταξή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στηρίζουμε τις προθέσεις της καινούργια ελληνικής κυβέρνησης να ε, ρήξη με τις πολιτικές προηγούμενης κυβέρνησης ε, και πιστεύουμε ότι έχει μια σημαντική ευκαιρία ε, να αναθεωρήσει τις παλιότερες πολιτικές σε ό,τι αφορά τη Μακεδονία. Συνεπώς καλωσορίζω τους, τις προσπάθειες να έρθουν οι Μακεδόνοι ηγέτες στο τραπέζι να διαπραγματευτούν αλλά αυτό δεν αρκεί πια η κυβέρνηση της Μακεδονίας θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως ε, μια πλήρως ε, διαφανή έρευνα για την τραγωδία του Κουμάνοβο και για τις ε, ε κατηγορίες περί παρακολουθήσεων. Αν δεν τα καταφέρουν θα πρέπει να αφήσουν την κυβέρνηση και να έρθει κάποιο άλλος να κυβερνήσει τη χώρα. Χρειάζεται πολλά να οικοδομηθούν στην πολιτική της Μακεδονίας και αυτό θα πρέπει να γίνει αμέσως. Uh, thank you. Uh, do you accept uh, blue card? Δέχεστε την μπλε κάρτα της κυρίας Ακοράφα; Please. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας θυμίσω κύριε συνάδελφε κάτι που είπαν οι πρέσβεις για την κυβέρνηση της Φύρομ μετά τη συνάντησή τους με τον κύριο Γκουρεύσκη έχουμε εκφράσει λένε τις ανησυχίες μας στον πρωθυπουργό ότι η κυβέρνηση δεν έχει σημειώσει πρόοδο σχετικά με τις σα σε περί κατάχρησης εξουσίας. αυτό δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσο η κυβέρνηση της χώρας είναι προσιλωμένη στις δημοκρατικές αρχές και αξίες της ευρωατλαντικής κοινότητας. η συνεχιζόμενη αποτυχία θα βλάψει την πρόοδο στην ευρωπαϊκή ένωση. Κύριε συνάδελφοι να ξεκαθαρίσουμε για μια ακόμη φορά ότι η ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της φύρομ με την προϋπόθεση ότι θα γίνονται σεβαστά τα κριτήρια της κοπενχάγης και θα σημειωθεί πρόοδος στις σχέση καλής γειτονίας. δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η φάρσα να ξεκινάμε διαπραγματεύσεις για χώρες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και οι κυβερνήσεις τους δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον να συμμορφωθούν με τις αρχές και τις αξίες της ευρωπαϊκής ένωσης. przypominam o limicie czasu na σας παρακαλώ πολύ να θυμάστε ότι υπάρχει και χρονικό όριο όταν έχετε ερώτηση με μπλε κάρτα, είναι 30 δευτερόλεπτα, μάξιμου. Παρακαλώ η απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ για την υπενθύμηση. Ε, ναι, συμφωνούμε πλήρως. Ε, εκτός από το γεγονός ότι δεν γίνονται διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Μακεδονίας αυτή τη στιγμή ακριβώς ε, επειδή η Ελλάδα τις μπλοκάρει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εκ μέρους του FDD, ο κύριος Μπάτεν. Ο κύριος Στελνίδης ε, Σκυλιανίδης πολύ καλά περιέγραψε την κατάσταση. Αναφέρθηκε στις βιότητες στο Βορρά. Μετά από μια μακρά πολιτική κρίση στη χώρα. Βέβαια η κατάσταση είναι πολύ πιο σοβαρή και φύση του προβλήματος. Έτσι δεν λύνονται τα συστηματικά προβλήματα. Η Επιτροπή πιστεύει ότι θα μπορέσει να διορθωθεί η κατάσταση εφόσον ε, είναι υποψήφια χώρα και ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 11 Μαρτίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την έκθεση πρόοδου για την ένταξη της ΦΥΡΟΜ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν άλλες πολλές χώρες δεν έχει σημασία φαίνεται πόση διαφθορά υπάρχει, πόσο μακριά βρίσκεται από τις απόψεις και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημασία έχει να ξαναμπεί, να μπει άλλη μια χώρα στη μεγάλη αυτή αυτοκρατορία. Ό,τι και αν λένε οι εμπειρογνώμονες, τους εύχομαι καλή τύχη. Ε, κύριος Ζαριανόπουλος οι επικίνδυνες εξελίξεις στη φύρομ και την ευρύτερη περιοχή δεν αποτελούν έκπληξη. είναι συνέπεια και συνέχεια της επέμβασης των ηνωμένων πολιτειών του νατο και της ευρωπαϊκής ένωσης στην περιοχή. η καλλιέργεια κρατικών μεγαλοδιατισμών και αλυτρωτισμών αξιοποιώντας το προτεκτοράτο του κωσυφοπεδίου εθνοτικών και θρησκευτικών διενέξεων η αλλαγή συνόρων η εναλλαγή αστικών κυβερνήσεων πατώντας τη λαϊκή δυσαρέσκεια για την αντεργατική πολιτική που ακολουθείται γίνονται εργαλεία για το ξαναμοίρασμα του πλούτου τον έλεγχο των δικτύων μεταφοράς στην περιοχή ιδιαίτερα της ενέργειας από επιχειρηματικούς ομίλους. τα δικά τους συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς τους με τα ρώσικα και αμερικάνικα μονοπόλια εξυπηρετούν και αποτυπώνουν οι εκθέσεις προόδου της ευρωπαϊκής ένωσης. οι λαοί της φύρων των βαλκανίων έζησαν ειρηνικά στον σοσιαλισμό στον καπιταλισμό γεύθηκαν βαρβαρότητα πόλεμο φτώχεια εκμετάλλευση. επιβάλλεται να είναι σε επαγρύπνηση για να ακυρώσουν τη συνέχιση των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων τα νέα δεινά που συνεπάγεται η ένταξη της φύρων και άλλων χωρών στην ευρωπαϊκή ένωση και τον νατο. Ευχαριστώ. Ε, Prime Minister ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Πέτρελ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, καταρχήν να ευχαριστήσω τον Επίτροπο τον κύριο Στυλιανίδη για τα πολύ σαφή λόγια του. Η Μακεδονία Φύρομ ε, ως υποψήφια χώρα περνάει από μια εσωτερική πολιτική κρίση και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις έχουν μπλοκαριστεί. Η χώρα έχει αποσταθεροποιηθεί πολιτικά και αυτό είναι σημαντικό και για την ίδια και για όλη την περιοχή. Ε, χαίρομαι για την έναρξη του πολιτικού διαλόγου ανάμεσα στη συμπολίτευση και την αντιπολίτευση συμπεριλαμβανομένων και των Μακεδόνων Αλβανών για προκειμένου να διευκολυνθεί η καλή λειτουργία του Κοινοβουλίου της χώρας και προκειμένου ο πολιτικός διάλογος να είναι υγιής. Ε, θέλω να συγχαρώ τους συναδέλφους που βοηθούν και ε, χαίρομαι που επικρατεί σοφροσύνη στο διάλογο. Η διαβούλευση είναι σημαντική γιατί θα πρέπει να λειτουργήσει πλήρως η κοινή κοινοβουλευτική επιτροπή, η μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή μετά από πολύ καιρό. Ε, προς όφελος της πολιτικής ε, σταθερότητας, της καλύτερης ε, γειτονίας και της ευρωπαϊκής προοπτικής θα πρέπει να πετύχουμε συγκεκριμένους και, συγκεκριμένη και απτή πρόοδο στην διαδικασία ένταξης της χώρας. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί μια ακόμα αιστεία ε, έντασης και κρίσης, ε, μια ακόμα σύγκρουση. Ε, υπάρχει, υπάρχουν ε, και διαθρησκευτικές αιτίες που μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιες κρίσεις, τέτοια κρίση. Νομίζω ότι αυτό είναι προς κοινό μας συμφέρον. ευχαριστώ. Μία μπλε κάρτα από τον κύριο Συναδεινό. Συναδινός. Συναδεινός. Κύριο Συναδεινός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο συνάδελφο που τους αποκαλεί Μακεδόνες, εγώ που κατάγομαι και γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Καστοριά, ένα νομό της Μακεδονίας, της Ελλάδος, πώς θα με αποκαλούσε ο κύριος συνάδελφος, Σκοπιανό. Mr. Prime Κύριε Πρωθυπουργέ, παρακαλώ. Ε, έχετε γεννηθεί, λέτε, στην Ελληνική Μακεδονία. Ε, οπότε δύσκολα μπορώ να φανταστώ ότι κανείς θα σε αποκαλούσε Σκοπιανό. Ο καθένας έχει την ταυτότητά του και πρέπει να μπορεί να ζει με βάση αυτή την ταυτότητα. Ο κύριος Φάλκενστάιν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον τελευταίο Βάγγελ, Κουκάνεν και Χάουτ και τον Επίτροπο για τις ε, διαπραγματευτικές τους ε, προσπάθειες. Ε, έχουν ένα δύσκολο καθήκον και αυτό το καθήκον είναι να καταλήξουν σε μια νέα αρχή χωρίς να ρίξουν ολόκληρη τη χώρα σε χάος ή ή χωρίς να επιτρέψουν ειρηνικές διαδηλώσεις να εκφυλιστούν και να εκτροχιαστούν σε βίες διαδηλώσεις. Ήμουνα στα Σκόπια την προηγούμενη εβδομάδα και είδα πόσες χιλιάδες ανθρώπων διαδήλωσαν για περισσότερη δημοκρατία, δικαιοσύνη, ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, για περισσότερες ενέργειες κατά της διαφθοράς και της εγκληματικότητας. Και το θέμα δεν είναι ότι μίλησαν σοσιαλδημοκράτες, πολύ σημαντικότερο ήταν ότι παρούσες ήταν πάρα πολλές, μια μεγάλη σειρά από ΜΚΟ, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Πολλοί άνθρωποι με διαφορετική εθνοτική προέλευση. Και όλα αυτά ήταν ειρηνικά, γιατί οι ε, διαδηλωτέ ήταν ειρηνικοί, αλλά να πω και ότι και η αστυνομία επέδειξε ευφυΐα. Αυτές λοιπόν οι εξελίξεις φέρνουν αυτή τη χώρα πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό πρέπει να το υποστηρίξουμε. Θέλουμε να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας ε, προς τους ε, φίλους και τις οικογένειές τους που έχασαν τη ζωή τους στο Κομάνοβο. Αλλά ξέρετε είμαι σίγουρος ότι εκεί δεν επρόκειτο για εθνοτική σύγκρουση αλλά για εγκληματικότητα. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε έτσι ώστε εμείς να μην βάλουμε το φυτίλι ωφέλη της εθνοτικής σύγκρουσης. Εύχομαι λοιπόν στους διαπραγματευτές μας επιτυχία και για να επιτευχθεί αυτή ε, πρέπει να υπάρχει και διάθεση συμβασμού. Αλλά μην αυταπατώμεθα. Κανένας ε, πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως ένας, ένας ίσως, αλλά εγώ τα έλεγα σχεδόν κανένας δεν θα μπορούσε να επιβιώσει αν αποκαλύπτοντο για τον ίδιο αυτά που αποκαλύφθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Για τον ίδιο και για την κυβέρνησή του. Κανείς δεν θα επιβίωνε. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του ECR, ο κύριος Νικολάη Παρέκοφ. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ως εκπρόσωπος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Ανησυχώ από τις προσπάθειες που γίνονται να κρατήσουμε όμοιρο τη χώρα αυτή εξαιτίας πολιτικών συμφερόντων. Ακόμα και ο Ρώσος υπουργό Λαυρόφ δήλωσε σήμερα ότι οι γείτονες χώρες θέλουν να μοιραστούν τη Μακεδονία. Δεν έχει νόημα. Η εθνοτική σύγκρουση το μόνο που κάνει είναι ότι έχει αρνητικές συνέπειες για όλη την περιοχή. Η μόνη λύση είναι ο ευρωπαϊκός δρόμος για τη χώρα αυτή, να διασφαλιστούν συγχρόνως τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Όμως τα δικαιώματα των, ε, της βουλγαρικής μειονότητας δεν τηρούνται. Συλληπιτήρια για όλους τους νεκρούς. Όμως εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βουλγαρικής προέλευσης απειλούνται σε μια χώρα η οποία βρίσκεται στο δρόμο προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς να δεχτούμε κάτι τέτοιο τη στιγμή που παραβιάζονται τόσα δικαιώματα. Ευχαριστούμε. Δέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Επιτίδιο. Yes, yes. Ναι. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε που αποδέχεστε την ερώτησή μου. Ε, είπατε προηγουμένως ότι πολιτικές σκοπιμότητες κρατούν όμοιρο την ε, χώρα της Φύρομ. Ήθελα να μου διευκρινίσετε την ερώτηση αυτή την απευθύνεται στην ηγεσία της χώρας η οποία όχι μόνο δεν πληρεί τα κριτήρια της Κοπεχάγης αλλά και δεν κάνει τίποτε προς αυτή την κατεύθυνση ή έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας. Μπορείτε να μου το διευκρινίσετε σας παρακαλώ αυτό. Please. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Είχα υπόψη μου τις συζητήσεις της Μακεδονίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι Βουλγάρος υπήκος, είμαι Ευρωβουλευτής τα τρία τέταρτα όμως των μελών της οικογένειάς μου έχουν γεννηθεί στη Μακεδονία. Είτε πρόκειται για το βουλγαρικό τμήμα είτε για το άλλο. Η χώρα αυτή θα έπρεπε να είναι ακέραια. Αυτό πιστεύω και δηλώνω ότι η Μακεδονία πρέπει να προστατεύει τα δικαιώματα όλων των ομοιονοτήτων και της βουλγαρικής. Ο κύριος Ράντος. Τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να σημειώσουμε ότι μετά τα δραματικά γεγονότα του Κουμάνοβο ε, δεν ακολούθησε, άλλη εθνο... δεν ακολούθησε εθνοτική σύγκρουση. Ε, έγιναν ε, διαμαρτυρίες, η κατάσταση ήταν πολύ έντονη, αλλά δεν επήλθε σύγκρουση, ε, η σύγκρουση. Αυτό σημαίνει ότι η Μακεδονία έχει οριμάσει. Βέβαια, για το θέμα αυτό θα πρέπει να επικριθούν οι αρχές, αλλά και το γεγονός ότι ε, οι ευρωπαϊκές προοπτικές ε, της Μακεδονίας δείχνουν να είναι πολύ ε, πιο πίσω από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια. Θα πρέπει η Μακεδονία να μπορέσει να δει καθαρά το ευρωπαϊκό της μέλλον. Ευχαριστώ τους κύριους Βάιτελ, Κούκαν και λοιπά που βοηθούν abgeordnete ε, ε, Vizepräsident Ulrike Lunacek, eine Minute bitte sehr. Η κυρία Λούνατσεκ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, νομίζω Όλοι μας ε, σοκαριστήκαμε από αυτή την βία επίθεση κατά των αθών πολιτών ε, στο Κουμάνοβο πριν από λίγες μέρες. Ε, είναι σαν να επανέρχονται τα φαντάσματα του παρελθόντος. Πρέπει λοιπόν να εξαστεί η όλη υπόθεση συμπεριλαμβανομένων και των υπονιών που υπάρχουν ότι ήταν δάχτυλο της κυβέρνησης Γκρουευσκή και των Ρώσων. Η κυβέρνηση δεν μπορεί βέβαια αυτό να το κάνει μόνη τη και αν όμως δεν κάνουν κάτι θα πρέπει η κυβέρνηση κυβέρνηση να Υπάρχουν δύο πράγματα που είναι σαφή. Ε, Σήμερα με τι δικέ μου ε, πληροφορίε, αυτή η επίθεση στο Κουμάνοβο ήταν καθαρά τρομοκρατική από επαγγελματίε, εγκληματίε ε, και δεν ήταν εθνοτική. Με μεγάλη χαρά είδα την προηγούμενη Κυριακή οι Αλβανοί και οι Σλαβομακεδόνε ε, διαδήλωσαν από κοινού στην Μακεδονία και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε. Και κάτι άλλο. Θέλω να απευθυνθώ στο ΕΛΚ να σταματήσει να υπερασπίζεται τους πολιτικούς της πολιτικής τους οικογένειας οι οποίοι απλά έχουν ξεφύγει τελείως από το δημοκρατικό δρόμο και από το κράτος δικαίου. Κυρία ε, Λούνατσεκ, δέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Κάρσκι. Παρακαλώ κύριε Κάρσκι, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής στην κυρία Λούνατσεκ. Ε, θα ήθελα να ε, πω ότι ε, αντιπροσωπεύω μια χώρα μικρή, όχι πολύ μακριά, ούτε πολύ κοντά στην Μακεδόνια. Τι πιστεύετε για το όνομα μια τέτοια χώρα. Είναι δύσκολο να ζήσει κανεί σε μια τέτοια χώρα και να ζήσει μια σταθερή ζωή ε, σε μια χώρα τη οποία το όνομα αμφισβητείται και δεν ξέρουν καν πώ ονομάζεται η χώρα του. Τι λέτε για αυτό το θέμα. Thank you, Mr. Karski, for the... Ευχαριστώ κύριε Κάσκι για αυτό το, αυτή την ερώτηση. Μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το θέμα το οποίο δεν πρόλαβα να συμπεριλάβω στην αρχική μου παρέμβαση στηρίζω όλους όσους καλούν την ελληνική κυβέρνηση, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ε, με την οποία εμείς συμπαθούμε ιδιαίτερα ως πολιτική ομάδα γιατί πολεμάει τη λιτότητα, πολεμάει, μάχεται προκειμένου να επιστρέψει η, κοινωνική ε, ειρήνη ε, στη χώρα κλπ. Νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να υποφεληθεί της ευκαιρίας για μια καινούργια αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μια συμφωνία για το όνομα της Μακεδονίας έτσι ώστε να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις η χώρα. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό κύριο Κοράου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κύριε Πρόεδρε, ε, βλέπουμε λοιπόν χτες τις διάφορες πλευρές που σαντήθηκαν αναζητώντας την διαβούλευση, πολύ δύσκολη διαβούλευση, ανάμεσα σε δύο μέρη τα οποία βρίσκονται σε αρκετά περίεργη πολιτική κατάσταση. Στη Μακεδονία έχουμε τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στους δρόμους, ένα κλίμα που γίνεται όλο και πιο εκρηκτικό. Νομίζω λοιπόν ότι εν μέρει αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας δεκαετίας που περιμένει η χώρα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί λοιπόν να γίνονται βήματα προς τα εμπρός, προς το κράτος δικαίου, γίνονται βήματα προς τα πίσω. Θεωρώ λοιπόν ότι εμείς έχουμε ευθύνες ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ευθύνες γιατί χάθηκε τόσος πολλής χρόνος και κυρίως ε, υπάρχουν συγκεκριμένα κράτη που έχουν πιο πολλές ευθύνες. Δράτω με τις ευκαιρίες ε, να στηρίξω αυτό που είπε η κυρία Λούρνατσοκ κυρίως απευθυνόμενη προς την ελληνική κυβέρνηση, την καλούμε πλέον να κάνει ένα βήμα σημαντικό προς τα εμπρός. Ο κύριος Συναδεινός παρακαλώ, έχει το λόγο. Το Δεκέμβριο του 2012 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι για να έχει ευρωπαϊκή προοπτική η φύρομ οφείλει να προωθήσει και να σεβαστεί τι σχέσει καλής γειτονίας, να εφαρμόσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσει και να συμβάλλει στην επίλυση του θέματος της ονομασίας υπό την αιγίδα του οηε. πιστεύει κάποιο σε αυτή την αίθουσα ότι οι έλληνες θα παραδώσουμε δυόμισι χιλιάδες χρόνια ιστορίας πολιτισμού και κληρονομιάς και θα συμφωνήσουμε στην ανεφόρον υπογραφή του πιστοποιητικού βάφτισης της φύρομ; πιστεύει κάποιος ότι αν τους ονομάσετε μακεδόνες θράκες σπαρτιάτες αθηναίους τότε πραγματικά αυτό το μόρφωμα κράτος έχει θέση στην ευρωπαϊκή ένωση; η φύρομ έχει ανοιχτά μέτωπα τόσο στο εξωτερικό αλλά κυρίως στο εσωτερικό. απλά ανατρέξτε στις εκθέσεις προόδου τη επιτροπής του οασέ αναρωτηθείτε γιατί η φύρομ βρίσκεται σε διένεξη με την ελλάδα τη βουλγαρία για ιστορικούς λόγους και την αλβανία για φυλετικούς μειονοτικούς λόγους. αναλογιστείτε αν το κουμάνοβο ή το τέτοβο παλιότερα είναι γεγονότα ίσονος σημασίας. ταξιδεύστε στον περλεπέ στην αγρίδα και στο μοναστήρι και μιλήστε περί μακεδονισμού. θα εκλαγείτε από τις απαντήσεις. είναι δύσκολο η ελλάδα να αποδέχεται στοικά τη συνεχή ύβρι ακόμα και από εκπροσώπους κρατών μελών της ευρωπαϊκής ενώσεως και τη συνεχή αναφορά τους στους κακούς έλληνες που αρνούνται την ευρωπαϊκή προοπτική της φύρομ. η αδιαλαξία και η αμετροέπεια έχουν κάποια όρια. ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ που δέχεστε την ε, μπλε κάρτα μου και την ερώτησή μου. Ε, πράγματι, δεν θα έπρεπε να, η συζήτηση να είναι φιλοσοφική, ποιο ε, πρέπει να είναι το όνομα, ποια, πώς λέγεται η περιοχή, πώς χωρίζεται η Μακεδονία κλπ. Μερικές χώρες έχουν αναγνωρίσει την Μακεδονία με το όνομα Μακεδονία. Το θέμα δημιουργήθηκε αργότερα ίσως. Ε, το θέμα όμως που πρέπει να μας απασχολεί είναι η περιφερειακή συνεργασία. Πρακτικά πράγματα, ε, τα οποία μπορούν να αλλάξουν μέσω των ημερών και πολυμερών σχέσεων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι τα πρακτικά βήματα τα οποία έχει λάβει για παράδειγμα η Ελλάδα τελευταία έτσι ώστε η Μακεδονία να ενταχθεί στην περιφερειακή συνεργασία και να βοηθηθεί να κάνει κάποιες μεταρρυθμίσεις που τόσο χρειάζονται. Ευχαριστώ. Αναπληρώτης δεν θα πρέπει η χώρα των Σκοπίων να εκφράζει αλυτρωτικές και επεκτατικές βλέψεις εναντίον άλλων χωρών, όπως είναι οι γειτονικές χώρες, η Βουλγαρία, η Αλβανία και η Ελλάδα. Ευχαριστώ. Christian Preda. Ο κύριος Πρέντα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συζητάμε εδώ και τη Μακεδονία και την προηγούμενη φορά έλεγα ότι ακόμα και αν πρόκειται για έκθεση πρόοδου σχετικά με τη χώρα αυτή, δυσκολευόμαστε να πούμε τη λέξη, γιατί πρόοδος, εγώ θα έλεγα ότι μάλλον ε, η κατάσταση πάει σημειωτών. και επιτόπου. Η πολιτική κρίση δημιουργεί νέες δυσκολίες. Στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε στη Μακεδονία είναι η απουσία νοτροπίας συμβιβασμού και πραγματικού διαλόγου. Εγώ χαιρετίζω, όπως και άλλοι συνάδελφοι, που οι τριμερείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βγάλει από τα διέξοδο την κατάσταση, από την άλλη μεριά η στρατηγική των ε, σοσιαλιστών βγαίνουν στους δρόμους για να αμφισβητήσουν την ε, ίδια την κυβέρνηση. Είναι δύσκολο και να διαπραγματευόμαστε από τη μια μεριά και να κατεβαίνουν στον δρόμο από την άλλη μεριά οι άνθρωποι. Χαίρομαι που κυρία Λούνατσε και άλλοι ενδιαφέρονται για τις σχέσεις του ΕΛΚ με το κράτος δικαίου κλπ. Αλλά θα ήθελα να δω την ίδια στάση και από πλευρά των σοσιαλιστών πρωθυπουργών στην Ευρώπη με κυβερνήσεις που όπως τη Ρουμανία έχουν καταδικασμένους υπουργούς. Ίσως να τα έχετε ακούσει. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να μην χρησιμοποιούμε το δρόμο για να διαλύουμε τους θεσμούς. Και δεν πρόκειται για το ΕΛΚ εδώ, πρόκειται για μια σοβαρή πολιτική κρίση. Και θέλω να προσθέσω, σε αντίθεση με του ελεύθερου σοσιαλιστέ κλπ., ότι υπάρχει και μια εθνοτική διάσταση σε αυτή την πολιτική κρίση που είναι πολύ επικίνδυνη. Δεν φτάνει εδώ να μιλάνε οι πράσινοι, οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλιστέ και να αρνούνται τη διάσταση αυτή. Είναι κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ανα πάσα στιγμή. Δέχεστε μπλε κάρτα από την κυρία Λούνατσεκ. Παρακαλώ κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρέντα, εμείς ως πράσινοι επικρίνουμε και τους σοσιαλιστές και το ΕΛ και μερικές φορές και τους ίδιους τους δικούς μας τις κυβερνήσεις όπου βρισκόνται. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Αυτό που εννοούσα είναι ότι αυτό το οποίο βλέπουμε και το είπαμε και χτες στη συζήτηση με τον κύριο Ορμπάν, αλλά τώρα έχει να κάνει με τον κύριο Γκρουεύσκη, ότι ορισμένοι από τη δικιά σας πολιτική οικογένεια είναι με το μέρος του παρόλο που έχει συμπεριφερθεί πολύ αυταρχικά τους τελευταίους μήνες και είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχετε υπόψη σας. Ευχαριστώ. Να απαντήσετε παρακαλώ, κύριε Πρέντα. Ναι, βεβαίως. Θα απαντήσω σε όλα αυτά. Εγώ δεν θέλω τη συζήτηση αυτή που έχει να κάνει με μια πολύ σοβαρή πολιτική κρίση σε μια χώρα, σημαντική για μας, να την κάνω συζήτηση για το ΕΛΚ. Η σωστή στάση για να βγούμε από τα διέξοδο δεν είναι να βρίσκουμε από δύο πεβαίους τράγους επειδή πολιτικά είσαστε πιο αδύναμοι και θέλετε να βρεθείτε εσείς οι πράσινοι στην ε, ατζέντα, στην πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια, δέχεστε και άλλη μια μπλε κάρτα από τον κύριο Νταμπάσκι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν πρόκειται για διαμάχη ανάμεσα στο ΕΛΚ, τους Πράσινους ή άλλο Ευρωπαϊκό Κόμμα. Πρόκειται για την ακαιρεότητα μιας βαλκανικής χώρας. Όσοι ζουν στα Βαλκάνια γνωρίζουν πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για μια εθνοτική σύγκρουση που είναι πολύ επικίνδυνη. Πρόκειται για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για διαφθορά. Συνεπώς, το πρόβλημα δεν έχει καμία σχέση με την διαμάχη δεξιάς και αριστεράς κύριε Πρέντα, να απαντήσετε. Συμφωνώ απόλυτα. Όντω πρέπει να επικεντρωθούμε στη Μακεδονία. Από την άλλη μεριά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι μπορούμε να κάνουμε και ζημιά ενθαρρύνοντας τα Βαλκάνια σε διάφορες βαλκανικές χώρες λύσεις οι οποίες δεν είναι παρά ιδεολογικές, ιδεολογικοί αυτοσχεδιασμοί. Έχουμε εξάλλου παραδείγματα στο πρόσφατο παρελθόν. Προσοχή λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Διαδικαστικό, ο κύριος Φουντούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έγινε κατάχρηση του θεσμού της μπλε κάρτας μεταξύ του κυρίου Πρέντα και της κυρία Λούνατσεκ. Δεν άκουσα καμία ερώτηση από την κυρία Λούνατσεκ, αλλά απλώς είχαν μια πολιτική αντιπαράθεση. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Ε, Deputy Sergei Stanishev, one and a half minute. Take a floor, please. Κύριο Στάνισεφ, 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Ε, πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, συνάλφη. Παλιότερα η Μακεδονία ήταν από τους, πρωτο, από χώρες για ένταξη εκ μέρους των χωρών Δυτικής, ε, των Δυτικών Βαλκανίων. Όμως, σήμερα περνάει μια πολύ βαθιά πολιτική κρίση και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πρόκειται για κάτι ευκαιριακό. Τα θέματα είναι θεμελιώδη που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε πώς καταφέραμε να φτάσουμε εδώ. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίμησε και υποβάθμισε αυτά που ελάμβαναν χώρα στην Μακεδονία για, πολύ καιρό. Μια κυβέρνηση η οποία θέσπισε ένα αυταρχικό καθεστώς που δεσπόζει στα μέσα ενημέρωση, στην οικονομία, ε, στη, στον τύπο και στη δικαιοσύνη την Κυριακή ήμουνα στις ε, διαμαρτυρίες ε, των πολιτών στη, στα Σκόπια. Δεν πήγα εκεί να κηρύξω, ε, ούτε να διδάξω. Πήγα για να ακούσω. Και είδα εκεί ανθρώπους διαφόρων εθνοτικών προελεύσεων, διαφόρων πολιτικών πεπιθήσεων, από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, από τα μέσα ενημέρωσης κλπ. Και όλοι ζητούσαν την εφαρμογή των δημοκρατικών αξιών. Ένας από τους ομιλητές από ένα φοιτητικό κίνημα, από το φοιτητικό κίνημα, ε, είπε δεν πρόκειται για την εξουσία αλλά για το πώς θα λειτουργεί το κράτος και αυτά τα γεγονότα δεν πρέπει να επαναληφθούν. Αυτά, αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στη στάση που θα κρατήσουμε σε ό,τι αφορά τη Μακεδονία. Γιατί η κρίση είναι βαθιά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνε. Ευχαριστώ. Э, Deputy Filis One minute. Take a please. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο και ο Μεστάνα του Φιλελεύθερου Κόμματος Βουλγαρία Βουλγαρίας ε, έστειλε μια επιστολή στην αρχή του χρόνου σε όλους τους ηγέτες, ε, τους ελεύθερους ηγέτες της Μακεδονίας και είπε, του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανοίξει ε, την αγκαλιά της στη Μακεδονία. Θα πρέπει να είμαστε εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δραστήριοι ε, για να εξασφαλίσουμε την ειρήνη και την ε, εδαφική ακαιρεότητα όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Η Μακεδονία πρέπει να ξεκινήσει το δρόμο που θα την οδηγήσει σε ευρωπαϊκές αξίες ε, και πρέπει να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα. Η Βουλγαρία έκανε μια ήπια μετάβαση από το απολυταρχικό καθεστώς προς τη δημοκρατία. Ελπίζω ε, ότι η Βουλγαρία μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Εσείς που είσαστε εδώ και κοιτάτε, βλέπετε λοιπόν πόσοι οι βουλευτές βρίσκονται εδώ ε, και ξέρετε πόσο κοστίζει αυτό το παιχνίδι και 250 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτή είναι η Ευρώπη της πατάλης, γιατί όσον αφορά την Φύρομ, γιατί Φύρομ λέγεται κύριοι και όχι Μακεδονία, γιατί Φύρομ λοιπόν θέλω να πω εξής, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται πάρα πολύ να μην περάσει από εκεί ο γογός του πετρελαίου και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκείνε οι οποίε ε, υποδαβλίζουν όλα αυτά τα κινήματα να μην περάσει ο αγωγό γιατί η η χώρα Φύρομ ε, έχει στραφεί προς τη Ρωσία γιατί η Φύρομ αναζητά διαφορετικές λύσεις. Δεν πιστεύετε λοιπόν ότι οι Αμερικανοί όπως κάνουν και σε ολόκληρο τον κόσμο θέλουν να βάλουν το δάχτυλό τους και όταν δεν τα καταφέρνουν είναι εκείνοι που υποδαβλίζουν ε, τις ομάδες για να επιτύχουν κάτι άλλο. Για σκεφτείτε λιγάκι κάπως καλύτερα, αντί να κοιμάστε όλη την ημέρα που κοιμάστε. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, ο κύριος Κοβάτσεφ, παρακαλώ. Μια στιγμή έκανα λάθος. Κύριε Μπονάνο, μπλε κάρτα από τον κύριο Νεκότιτς. Δέχεστε? Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, κύριε Μπονάνο που δεχτήκατε την μπλε κάρτα μου. Ε, ε, δεν μπορώ να κάθομαι εδώ χωρίς να αντιδρώ πια. Ε, ήρθα σε 9 το πρωί ε, και κάθομαι εδώ από τότε. ο πρόεδρος σας ήρθε εδώ και μίλησε για τη μετανάστευση και το πρώτο που είπε ότι είναι ότι η αίθουσα είναι άδεια παρόλο ότι η συζήτηση είναι πολύ σημαντική. Και μόλις τελείωσε, σκόθηκε και έφυγε. Ε, νομίζω ότι είναι υποκριτικό. To nie było pytanie. Bardzo proszę. Next blue card. Do you accept? Ε, και άλλη μια μπλε κάρτα. Δέχεστε. Mr. Polchak, take a floor, please. Κύριος Polchak. Thank you, Mr. President. Uh, thank you for accepting the blue card. Ευχαριστώ πολύ που δέχεστε την μπλε κάρτα μου. Η ερώτησή μου είναι πολύ απλή και σύντομη. Ε, εσείς μένετε εδώ συνέχεια, δεν φεύγετε ποτέ. Eh, λοιπόν, κοιτάξτε, πριν σας πω τη δική μου την ιστορία, να σας πω ότι εγώ είμαι και δήμαρχος στην Ιταλία και εκλέγομαι για 21 συναπτά έτη. Και θέλω να σας πω ότι αν δείτε τα δικά μου ποσοστά ψήφων και το τι κάνω, ε, θα πρέπει να είμαι στους πρώτους 50 των βουλευτών ε, που έχουν αυτή την αποδοχή. Επειδή λοιπόν είμαι κάποιος που τα λέω κατάμουτρα, σας λέω αυτό που σκέφτομαι. Ε, μερικές φορές μιλάω και άσχημα, χρησιμοποιώ ύβρις, αλλά προσπαθώ να υβρίζω παρά να είμαι υποκριτής όπως πολλοί από εσά. Όχι όλοι, αλλά πολλοί. Τι κάνουν πολλοί, γελάνε, κάνουν αστιάκια και σκασίλα τους για τον ευρωπαϊκό Λόγο. Το καταλάβατε? Uh, Ευχαριστούμε. Τώρα, σίγουρα πια ο κύριος Κόβατσεφ. Έτσι, μισή λεπτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, Οι πολιτικές ελίτ της Μακεδονίας πρέπει πάση θυσία να λύσουν την κρίση και να παραιτηθούν από κάθε σύγκρουση και κάθε διαμάχη. Όμως, λυπούμεθα που ο Πρωθυπουργός Γκρέσκι απομάκρυνε από τον ευρωπαϊκό δρόμο τη χώρα. Δεν βλέπουμε κανένα σημάδι καλής θέλησης υπερδημοκρατικών πρακτικών, η ισοτιμίας μεταξύ των πολιτών. Αντίθετα, οι σχέσεις με τις γείτονες χώρες έχουν επιδεινωθεί. Οι πρακτικές, οι παλιές, οι ολοκληρωτικές εξακολουθούν να παραμένουν. Και η επιθετική στάση επίσης για μια νέα ταυτότητα. Είναι λοιπόν προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Μακεδονία να είναι σταθερή και δημοκρατική χώρα με ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και να τηρούνται το δίκαιο και τα δικαιώματα. Οι θέσεις της Μακεδονίας όμως είναι κάπως περίεργες. Ο Υπουργός Λαυρόφ αναφέρθηκε σε κατακαιρματισμό της Μακεδονίας στις γείτονες χώρες. Οι πολίτες της Μακεδονίας δικαιούνται με διαφάνεια κυβέρνηση και δημοκρατική και δεν μπορεί να κρατούνται όμοιροι για να μπορεί να επιβιώσει ένας πολιτικός ηγέτης ο οποίος προσπαθεί να φανεί σαν εκείνος που θα σώσει. Ε, δέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Σάμι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συμφωνώ μαζί σας για κάποια θέματα. Έχω όμως και ένα πρόβλημα σοβαρό. Έχω μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι είναι φυσιολογικό να λέμε ότι φταίει για όλα η Μακεδονία ενώ τα δικά μας θεσμικά όργανα δεν βοηθούν αρκετά τη Μακεδονία και αποσταθεροποιούμε τη χώρα και την κάνουμε να πιστεύει ότι δεν μπορεί να προσεγγίσει στην Ευρώπη. Την ευθύνη λοιπόν να μην τη ρίχνουμε μόνο στη Μακεδονία. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα Βαλκάνια ήταν πάντα μια προβληματική περιοχή. Σας ζητώ λοιπόν για άλλη μια φορά, πιστεύετε ότι για όλα αυτά η Μακεδονία και μόνο. Απάντηση. Παρακαλώ. Ναι, βέβαια, αγαπητέ συνάδελφε, η ευθύνη είναι διπλή και η αλληλεγγύη πρέπει να γίνει αποδεκτή η χείρα βοηθείας. Όμως είναι ανεξάρτητη εδώ και 25 χρόνια περίπου η χώρα. Η Μακεδονία δεν μπόρεσε να έχει καλές σχέσεις με τους γειτονές της και δεν καταφέρνει να αποδείξει ότι πραγματικά θέλει καλές σχέσεις. Δεν έχει δείξει αυτή την καλή βούληση η Μακεδονία θέλει μια ταυτότητα η οποία δεν έχει ιστορικές ρίζες, δεν έχει ιστορικές αποδείξεις. Είναι προφανές λοιπόν ότι υπάρχουν συγκρούσεις. Το να χειραγωγούμε το παρελθόν είναι κακό για το μέλλον. Όμως έχουμε κάνει συστάσεις στις εκθέσεις μας, αλλά η Μακεδονία δεν τις εισακούει. Ευχαριστούμε κύριο Σπικουλέ, ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ πολύ. Η Μακεδονία γεωγραφικά είναι μια μικρή χώρα, όμως αποτελεί τμήμα μιας πολυτάραχης ε, περιοχής. Την Μακεδονία την ε, βλέπουμε πολύ συχνά μόνο υπό το πρίσμα των προβλημάτων με το όνομά της σε σχέση με την Ελλάδα. Όμως υπάρχουν και άλλα προβλήματα, η τρομοκρατία, η παρακολουθήση των πολιτών, η διαφθορά που πολύ συχνά μας ξεφεύγουν. Ε, επίσης, ο ισχυρός κομματισμός, επίσης, ε, ο πολιτικός διάλογος είναι ευκταίος, αλλά δεν λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή. Η χώρα αυτή ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της πορεία πριν την Κροατία, αλλά ακόμα βρίσκεται πάρα πολύ μακριά. Όλοι θα πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους για αυτή την κατάσταση και να προσπαθήσουν να βρουν μια πολιτική λύση το συντομότερο δυνατό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει. Ευχαριστώ. E, η κυρία Άννα Ζαμπόσκα. Δύο λεπτά παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Μακεδονία εδώ και δέκα χρόνια περιμένει να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μέρος της ευθύνη για την κλιμάκωση της βίας μετά τις εκλογές που έγιναν πέρυσι. Οι παρατηρητές στις εκλογές δεν διαπίστωσαν ελλείψεις κατά τη διάρκεια των εκλογών αυτών, όμως οι δηλώσεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπής καθώς και ορισμένων χωρών μελών είναι, ε, αποτέλεσαν μια ένα στοιχείο για τους κομμουνιστές να αρνηθούν την εντολή τους η πρέσβυρα των κάτω χωρών, για παράδειγμα, αναφέρθηκε σε έλλειψη συμφωνίας για τις δράσεις των πολιτικών κατά τη διάρκεια των εκλογών και το κατέδειξε ως πρόβλημα. Μπορούμε λοιπόν να αφισβητήσουμε στη μισή χώρα τα αποτελέσματα των εκλογών στις μισές χώρες με αυτόν τον τρόπο. Εγώ επισκέφθηκα τη χώρα και παρά τη βαθιά κρίση εξακολουθεί να είναι δημοκρατική χώρα η Μακεδονία που έχει τη θέση τη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνω έκκληση λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αρχίσει τι διαπραγματεύσει προσχώρηση με τη χώρα αυτή χωρί προκαταλήψει. Κάνω έκκληση επίση στου πολιτικού και στου κατοικού τη χώρα για να λυθεί το πρόβλημα όσον αφορά το όνομα αυτή τη νέα δημοκρατία. Η σταθερότητα στα Βαλκάνια είναι προ το συμφέρον όλων μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Πλένκοβιτς. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας θα ήθελα να υποστηρίξω την Μακεδονία και την ε, πορεία της προς την Ευρώπη. Κατά κάποιο τρόπο ε, είμαστε γείτονες της Μακεδονίας. Εγώ προέρχομαι από την Κροατία και ε, ένα τμήμα της δικής μας ευρωπαϊκής πορείας ήταν παράλληλο με, αυτό, με αυτήν της Μακεδονίας η, η Μακεδονία υπέγραψε το 2000 τη Συμφωνία Σύνδεσης και 15 χρόνια μετά δεν έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το γεγονός νομίζω συνεισέφερε στα δυσάρεστα γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από δύο εβδομάδες. Ε, η αντιπολίτευση δεν πρέπει να μπλοκάρει την λειτουργία του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να επιστρέψει το Κοινοβούλιο και η κυβέρνηση από τη μεριά της θα πρέπει να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για όλα τα δεινά η κοινή προσπάθεια του Επιτρόπου κ. Χάν και η δική μας πιστεύω θα πρέπει να βοηθήσουν, να βοηθήσουν στην χώρα να αποφύγει στο μέλλον γεγονότα όπως αυτά το Κουμάνοβο και ε, ελπίζουμε ότι οι Αλβανοί της Μακεδονίας ε, δεν θα πέσουν στην ε, παγίδα αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βέρ, ένα λεπτό. Ένα κράτος το οποίο εδώ και μια δεκαετία αναπτύσσεται αρκετά γρήγορα αντιμετωπίζει σήμερα μια κρίση και οι λόγοι είναι δύο. Πολιτική καταρχήν. Ε, η κυβέρνηση ε, κατηγορείται ε, για παρακολουθήσεις και άλλες παράτυπες δραστηριότητες. Ε, το έχουμε δει στο παρελθόν αυτό και στη Σλοβενία και στην ε, Βουλγαρία για να μην πω και στη Σλοβενία ε, οι τρομοκρατικές πράξεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εθνοτικές διαταραχές είναι επικίνδυνο. Θα πρέπει το πρόβλημα να λυθεί με την ένταξη της ε, χώρας ε, όσο το πιο γρήγορα γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν γίνει αυτό η κατάσταση νομίζω θα είναι πολύ πιο σταθερή. Δεν θέλουμε να γίνει θύμα ε, διαφορετικών και ξένων συμφερόντων αυτή η χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σπυράκη έχει τώρα το λόγο. Ένα λεπτό κύριε πρόεδρε κύριε επίτροπε το γεγονός ότι η πρώην ιουγκοσλαβική δημοκρατία της μακεδονίας είναι ευάλωτη σε επεισόδια όπως αυτά στο κουμάνοβο αναδεικνύει ότι στη χώρα υπάρχει σοβαρό έλλειμμα στη λειτουργία της δημοκρατίας. η κυβέρνηση της πρώην ιουγκοσλαβικής δημοκρατίας της μακεδονίας δεν σέβεται τη συμφωνία της αχρίδας και άρα τα δικαιώματα της πολύ ισχυρή σε σχέση με τον τοπικό πληθυσμό αλβανικής μειονότητας αλλά δεν είναι μόνο αυτό η αντιπολίτευση δεν κάθεται στα έδρανα της βουλής στα σκόπια από την ώρα που έγιναν εκλογές η κυβέρνηση δεν έχει πείσει ότι διενεργείται ανεξάρτητη έρευνα για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στις οποίες παρεμπιπτόντως πρωταγωνιστεί ο εξάδελφος του πρωθυπουργού Γκρούευσκι, ο οποίος βρίσκεται μάλιστα και εδώ στο στρασβούργο συνοδεύει τον πρωθυπουργό σύμφωνα με τον τύπο ο πρωθυπουργό γκρούευση μιλά για ξένο δάχτυλο στην πολιτική ζωή της χώρας την ώρα που η ρωσία δια του σεργέη Λαυρόφ, βλέπει πίσω από την αναταραχή που προκάλεσαν οι υποκλοπές προσπάθεια να αποτραπεί η συμμετοχή των σκοπίων στον turkish stream όλα αυτά είναι σενάρια συνωμοσία ενώ είναι φανερό ότι δεν υπάρχει σεβασμό των δικαιωμάτων όχι μόνο των αλβανών αλλά και των ρωμά και οι ελευθερίε του τύπου καταστρατηγούνται. έχουμε ευθύνη να κάνουμε συστάσει στι υποψήφιε χώρε στην περιοχή με πρώτη την πρώην γιουγκοσλαβική δημοκρατία τη μακεδονία ώστε να πέσει η ένταση και αλήθεια μετά από όλα αυτά πιστεύει κανένας εδώ ότι το μοναδικό εμπόδιο για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις της πρώην ιουγκοσλαβικής δημοκρατίας της μακεδονίας με την ευρωπαϊκή ένωση είναι η διαφορά τους με την ελλάδα; θέλουμε στα αλήθεια να ανοίξουμε την πόρτα της ένωσης σε μια χώρα που καταστρατηγεί βασικές αρχές στη λειτουργία της δημοκρατίας; σας ευχαριστώ. Η κυρία Πέτυρ. Ενάμιση λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των αστυνομικών της Μακεδονίας που έχασαν τη ζωή τους στο Κουμάνοβο. Ελπίζω ότι όσοι βρίσκονται πίσω από τις βάρβαρες αυτές πράξεις θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν και θα ληφθούν μέτρα για να αποφύγουμε τέτοια επεισόδια στο μέλλον. Εάν η Μακεδονία είχε ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αντί να τις βάζουμε εμπόδια, τότε τέτοια τυχή γεγονότα δεν θα είχαν λάβει χώρα. Και λυπάμαι που βλέπω πως η κατάσταση δεν κάνει την αντιπολίτευση να αλλάζει γνώμη και να βοηθήσει να βρεθούν λύσεις στο Κοινοβούλιο υπέρ του Μακεδονικού λαού. Όμως ποιος φταίει για την τραγική αυτή κατάσταση στη Μακεδονία. Στην πραγματικότητα ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο, γιατί ανεξάρτητα από όλα τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για άλλη μια φορά βάζει εμπόδια στο δρόμο της Μακεδονίας προκειμένου να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τη χώρα αυτή. Αν είχαν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είχαμε τέτοιε απόπειρε αρπαγής της εξουσίας μετά τις εκλογές και ούτε τέτοια προβλήματα με την κυριαρχία της χώρας. Για άλλη μια φορά το λέω. Έχει τηρήσει τι προποθέσει όλε η χώρα και πρέπει να με την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Τα διμερεί προβλήματα για το όνομα πρέπει να λυθούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Είχαμε και το παράδειγμα με την Κροατία και τη Σλοβανία, πέτυχε η διαδικασία εκεί. Η σταθερότητα τη Μακεδονία είναι πολύ σημαντική για τη σταθερότητα ολόκληρη τη περιοχή και τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Περνάμε στη διαδικασία Catch the τώρα. Ο κύριος Κύρτσος. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν τέσσερι βασικέ προποθέσει για να αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη συνεργασία τη με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονία και να ανοίξει ο δρόμο για μια μελλοντική ένταξη. Πρώτον, πρέπει να εκδημοκρατιστεί το πολιτικό σύστημα, το οποίο έχει αυταρχικά χαρακτηριστικά. Δεύτερον, πρέπει να σταματήσει η κυριαρχία του οργανωμένου εγκλήματο και των παρακρατικών ομάδων. Τρίτον, πρέπει να υπάρξει σεβασμό τη αλβανόφωνης μειονότητα τη χώρα για να αποτραπεί η επανάληψη του εμφυλίου. τέταρτον πρέπει να λυθεί το ζήτημα τη ονομασία με έναν έντιμο συμβιβασμό που θα ικανοποιεί τόσο τα σκόπια όσο και την αθήνα. επειδή είμαι Έλληνα και μπορεί να θεωρήσετε ότι δίνω αποκλειστική σημασία στο τέταρτο σημείο καλώ αυτού που ασκούν εξουσία στα σκόπια να ξεκινήσουν τη μακρά ευρωπαϊκή του πορεία βελτιώνοντα την κατάσταση στα τρία πρώτα ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μαδάμ Ρούζα Τόμασιτς. Κυρία Τόμασιτς. Καλή stanje u η τρέχουσα κατάσταση στη Μακεδονία είναι πραγματικά ανησυχητική, η κυβέρνηση είναι ασταθής, υπάρχει εθνοτική ένταση, δεν επικρατεί κράτος δικαίου, με άλλα λόγια είναι αδύνατο να εξασφαλιστεί ε, η οικονομική ευημερία, Εντάξει, ο λαός ε, είναι όλο και πιο ε, δυσαρεστημένος και βγαίνει στους δρόμους ευρωπαϊκή πορεία της χώρας είναι μπλοκαρισμένη, οπότε δεν υπάρχει και πολλή ελπίδα. Ε, η χώρα μπορεί να γλιστρήσει στην Άβυσσο και θα πρέπει να το αποφύγουμε, να το προλάβουμε. Οι υπηρεσίες, ε, μυστικές υπηρεσίες της Μακεδονίας, ε, από ό,τι φαίνεται, κάνουν τα δικά τους και αυτό καθιστά τη χώρα πριν τη ε, δεν θα πρέπει να περιμένουμε να ανάψει φωτιά. Ευχαριστώ. Take a floor, please. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, το πρόβλημα της ε, Μακεδονίας δεν είναι μακεδονικό. Είναι βαλκανικό και είναι και πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μακεδονία ήταν απομονωμένη για αρκετά χρόνια και αυτό είναι ένας από τους λόγους, μια από τις της ε, σημερινής κρίσης. Θα πρέπει καταρχήν να επιλύσουμε τα διμερεί προβλήματα, γιατί αλλιώς η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα γίνει δυνατή. Θα ήθελα επίσης να πω ότι στα Βαλκάνια Υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να λυθούν πριν την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κατόπιν της ένταξης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την, ε, πολιτεία των, για την κοινωνία των πολιτών σε νέες δημοκρατίες όπως αυτή της Μακεδονίας. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε αυτές τις ε, χώρες σε ένα λίμπο, σε μια ουδετερότητα ε, στο σύνολο μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Θα πρέπει επίσης να προλάβουμε την ριζοσπαστικοποίηση της κοινωνίας. Γι' αυτό το λόγο στην αρχές, στις αρχές Σεπτεμβρίου θα διοργανώσουμε ένα συνέδριο για να συζητήσουμε τη νέα στρατηγική για την περιοχή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χρυσόγονος. Πολλοί ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν στο ζήτημα της ονομασίας της ΦΥΡΟΜ και στη διαφορά με την Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά έχουν επιδείξει ετοιμότητα συμβιβασμού στο θέμα αυτό και το έχουν δηλώσει άλλωστε. το πρόβλημα προέρχεται από την άλλη πλευρά προέρχεται από αυτό που είπε ακριβώς ο ευρωβουλευτής του ευρωπαϊκού λαϊκού κόμματος ο κύριος πρέντα ότι δεν υπάρχει νοοτροπία συμβιβασμού εκ μέρους του πολιτικού συστήματος των σκοπίων και ειδικότερα εκ μέρους της κυβέρνησης γκουρεύσκη η οποία με τον τρόπο αυτό με τον αποπροσανατολισμό του λαού της σε θέματα παροχημένα όπως είναι θέματα εδαφικών διεκδικήσεων τα οποία κατ' ουσίαν υποκρύπτονται κάτω από το ζήτημα της ονομασίας θέλει να ε, τραβήξει την προσοχή του λαού από τα τρέχοντα προβλήματα στα οποία επιδεικνύει και ε, εντελώς αυταρχική διάθεση. συνεπώς το ζήτημα βρίσκεται από εκείνη την πλευρά και όχι από την πλευρά της ελλάδος. Ε, ευχαριστώ. Ε, Δέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Μάνες. Από τον κύριο Μαριά. Πρόεδρε, δεν ζήτησα μπλε κάρτα. Ήθελα να σας επισημάνω διαδικαστικά το εξής. Ότι έχουν δοθεί πάρα πολλές μπλε κάρτες. Εμείς περιμένουμε εδώ για το Catch the Eye. Ήμουν από τους πρώτους που ζήτησα Catch the Eye. Και αν συνεχιστεί αυτή η διαδικασία είναι λάθος. Να προτείνω λοιπόν. Πρώτον, όσοι είναι ομιλητές να μην κάνουν μπλε κάρτα διότι μιλούν δυο φορές και όσοι κάνουν μπλε κάρτα να μην μπορούν να μπουν στο catch the eye. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μιλούμε όλοι. Αυτό σας επέδειξα άτυπα. Δεν θέλω να κάνω ερώτηση στον συνάδελφο. Ε, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συμβουλή. Ο κ. Σόλτας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συνάδελφοι, η Μακεδονία βρίσκεται σε μια πολύ δυσχερή συγκυρία. Πριν από μερικούς μήνες ακόμα μιλούσαμε για τη Μακεδονία και την ευρωπαϊκή της ε, πορεία ή την πορεία εντάξει στο ΝΑΤΟ. Τώρα πια έχουμε καταλάβει ότι η ειρήνη είναι ε, πολύ ευπαθές ε, υλικό. Ε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην Μακεδονία. Ο χρόνος θα το δείξει. Ο χρόνος θα δείξει την σημασία εξωτερικών παραγόντων που προσπαθούν να επηρεάσουν τη γεωστρατηγική θέση της χώρας. Όμως, είναι αλήθεια ότι η Μακεδονία έχει πλέον καταστεί δαποθήκη. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσπαθήσουμε και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βάγκελ και την ομάδα του για τις ε, προσπάθειές τους. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουν προς την ίδια κατεύθυνση και ότι θα πετύχουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Πάιτ. Ο Υπουργός Πάιτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πριν από δέκα χρόνια η Μακεδονία ήταν μια χώρα των Δυτικών Βαλκανίων που πλησίαζε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Και τελικά τις κλείσαμε την πόρτα. Δεν έχουν ανοίξει οι διαπραγματεύσεις, δεν έχουν αρχίσει. Η χώρα, ειλικρινά, έχει χάσει τη διάθεσή της γιατί βλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε συνομιλίε. Τι νομίζετε λοιπόν, όλες αυτές οι αρνητικές απαντήσεις που έχει πάρει η Μακεδονία, τι νομίζετε εσεί, νομίζετε, δεν νομίζετε ότι έχει επηρεάσει τις εξελίξεις στη χώρα. Ευχαριστώ. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Είναι σωστή δικαιολογημένη η ερώτησή σας και κάποιες απαντήσεις ακούσαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι η προβληματική αυτή των σχέσεων της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν παρελθόν. Η Μακεδονία αποτελεί μέρος της περιοχής αυτής όπου η σταθερότητα και η ειρήνη είναι ευάλωτε. Όπως και να έχουν τα πράγματα πάντως, κάποιες δραστηριότητες πρέπει να αναλυθούν έγκαιρα προκειμένου να αποφύγουμε τέτοιου είδους δυσκολίες στο μέλλον όπως είδαμε τις τελευταίες μέρες στη Μακεδονία. Θέλω να ενημερώσω τους ευρωβουλευτές ότι σύμφωνα με τη διαδικασία Catch the Eye έδωσα το λόγο στους ευρωβουλευτές που δεν συμμετείχαν στη συζήτηση προηγουμένως και δεν ζήτησαν μπλε κάρτα. Τώρα λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από τον Επίτροπο να πάρει το λόγο εκ μέρους της υπατοεκπροσώπου. Please. Micro. Ήρθα εδώ για τη συζήτηση και βρίσκω πολύ απογοητευτικό όπως και ο Έλληνας συνάδελφος Μία μπλε κάρτα, δύο μπλε κάρτε επιτρέψατε που δεν ήταν καν ερωτήσει πολλέ φορέ. Δώσατε μπλε κάρτε και στο Κατστιάι. Ενώ ο προηγούμενο πρόεδρο είπε ότι δεν επιτρέπεται. Και κλείνετε τώρα τη συζήτηση. Κανένα δεν θα θέλει να έρχεται εδώ, άμα δεν παίρνουμε το λόγο. Ήρθε εδώ, όπω και ο συνάδελφο πριν, καλή την πίστη να ακούσω τη συζήτηση, σήκωσα το χέρι μου για το Catch και κάτω από τις προϋποθέσεις που μόλις αναφέρατε έπρεπε να μου έχετε δώσει το λόγο. Δεν μου το δώσατε όμως. Γιατί, τι συμβαίνει. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας κύριε. Όπως διαπιστώσατε έδωσα το λόγο σε έναν από κάθε πολιτική ομάδα. Αν υπάρχουν ευρωβουλευτές οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι με τη διεξαγωγή της συζήτησης, λυπούμε ειλικρινά. Και ελπίζω να τα καταφέρω καλύτερα την επόμενη φορά. Κύριε επίτροπε έχετε το λόγο. Ε, Ακούστε. Η συζήτηση έκλεισε. Και δίνω το λόγο στον Επίτροπο. Κύριε Επίτροπο, έχετε το λόγο. Γιατί δεν μου επιτρέπετε να... Με επιτρέψετε προηγούμενα στον άλλο. Γιατί δεν επιτρέπετε σε μένα. Επιτέλους σεβαστείτε με 93 ε, χρονών και είμαι από το πρωί εδώ. Σεβαστείτε το επιτέλους. Ja bardzo, panie pośle, bardzo pana szanuję osobiście, e, ale... Ακούστε κύριε, σέβομαι πάρα πολύ το άτομό σας αλλά ακολουθώ τις διαδικασίες. Αυτές με περιορίζουν. Δίνω το λόγο στον Επίτροπο. Θα ήθελα ο Επίτροπος να πάρει το λόγο. Μένουμε πίσω στο χρόνο. Ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ. Έχουμε κάποιους κανόνες και πρέπει να τους τηρούμε. κάνει παραβίαση. Nie, ναι, panie ε, ε, Υπάρχουν κάποιοι κανόνες και κάποιες διαδικασίες που καθορίζονται από τον κανονισμό και πρέπει να τους τηρώ. Σας παρακαλώ λοιπόν και εσείς να τηρείτε τους κανονισμούς. Και δεν με αφήνετε να την Την παραβίαση θέλω να πω. Λυπάμαι κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πολιτική πρωτοβουλία της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, όπως είπαμε. Πρέπει να προασπίσουμε μια επικοδομητική προσέγγιση από όλες τις πλευρές. Έτσι ώστε αυτή η πρωτοβουλία να πετύχει το στόχο της. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Η Αντιπρόεδρος κυρία Μογκερίνη και ο Επίτροπος κ. Χάν ε, θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση από κοντά και σίγουρα θα σας ενημερώσουν για περαιτέρω εξέλιξεις. Είμαι σίγουρος θα το κάνουν. Είδαμε μια συζήτηση με πολλές κόντρες αλλά και πολύ επικοδομητική. Όλοι μας ευχόμαστε το αποτέλεσμα να είναι συγκεκριμένο και η πρωτοβουλία αυτή να δώσει, να έχει συγκεκριμένη έκβαση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Ε, chciałem tylko Τώρα, θα ήθελα να υπενθυμίσω στους ευρωβουλευτές ότι ο 142.12 λέει ότι όσοι ευρωβουλευτές δεν συμμετείχαν σε μία συζήτηση μπορούν να υποβάλουν γραπτή δήλωση μέχρι 200 λέξεις που θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά της συζήτησης. Καλό λοιπόν τους ευρωβουλευτές που δεν είχαν την ευκαιρία να πάρουν το λόγο να το κάνουν. Τώρα, τελειώνουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό και δίνω το λόγο στο συνάδελφο.